λάβουμε υπόψη το ότι ολοένα και ε, πιο περίπλοκες είναι οι μέθοδοι ε, παραποίησης και πλαστογραφίας, οπότε και εμείς θα πρέπει με τη σειρά μας να καταπολεμήσουμε ε, αυτές τις πράξεις. Και μας απασχολεί, μας προβληματίζει το τι γίνεται στα σύνορα. Εμείς ακόμα δεν έχουμε μπει στο Σέγγελ, ελπίζω να μπούμε σύντομα, αλλά θέλω να εξασφαλίσω την ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων. Και αυτό μπορεί να γίνει και με το εν λόγω σύστημα. Αλλιώ να βρούμε και άλλα συστήματα. Ζόντσα. Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με το σχέδιο κειμένου και θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια πήγε πολύ καλά και θεωρώ ότι η ασφάλεια είναι το πιο κοινό από τα θέματα που μας απασχολούν. Είμαστε υπέρ του φάντο, αλλά πρέπει να θωρακίσουμε και την Frontex, γιατί είναι μια υπηρεσία με τεράστια σημασία. Θα πρέπει να είναι ολοένα και πιο αποδοτική για την ασφάλεια της Ευρώπης. Έχουμε πολλές αρνητικές εμπειρίες σε σχέση με την ε, παραβίαση των κανόνων της ε, ασφαλείας. Οπότε τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει κάποια βήματα προς την ασφάλεια. Αυτό κάνει και η Πολωνία. Άρα θα πρέπει να είναι εξίσου ασφαλής και η Ευρώπη. Αυτό κάνει και αυτό που τα κατά την αυτή η πρόταση. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε και τώρα. Το λόγο έχει η κυρία Ντάλι, η Επίτροπος Ντάλι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ για τη δουλειά σας, κυρία Μετσόλα, και ευχαριστώ και όλους τους ευρωβουλευτές για τη συζήτηση. Όπως προείπα, το ΦΑΝΤΟ θα βοηθήσει να έχουμε ένα υψηλό επίπεδο ασφαλεία εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενισχύσουμε του ελέγχου στα εξωτερικά μα σύνορα. Η τελική πολιτική συμφωνία για την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει σοβαρές βελτιώσεις, προσφέρει σοβαρές βελτιώσεις στο υπάρχον σύστημα και επιτρέπει να καταπολεμήσουμε την επεξαίρεση ταυτότητας, την κλοπή ταυτότητας και την διακίνηση πλαστών εγγράφων. Όπως είπαν πολλοί βουλευτές, θα έχουμε ένα ευρωστότερο σύστημα προστασίας των εγγράφων και των δικαιωμάτων των πολιτών. Υπό το φως της συζήτησή σας αναμένω την υπερψήφιση της τελικής συμβαστικής πρότασης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Μετσόλα, για την τελική της παρέμβαση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και πάλι σας ευχαριστώ, Επίτροπε Ντάλη. Παρακολούθησα με ιδιαίτερη προσοχή όλες τις παρεμβάσεις και θέλω να ευχαριστήσω για την ομόφωνη την αμέριστη στήριξη προς την έκθεση αυτή. Να θυμηθούμε ξανά για το τι μιλάμε εδώ. Το ΦΑΝΤΟ ε, είναι ένα σύστημα που θέλει να υποστηρίξει τις αρχές των 100 μελών στην ανταλλαγή, την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών. Επίσης την σωστή διάκριση γνησίων και πλαστών εγγράφων η χρήση πλαστών εγγράφων στην περιοχή, στον χώρο του Σέγγεν, έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, ιδίως τα πιο πρόσφατα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να αναλάβουμε δράση. Αλλάζει βεβαίω η μέθοδο τη ε, παραχάραξη των εγγράφων, γι' αυτό θα πρέπει να μπορούμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά σε σχέση με όσου θέλουν να παρανομήσουν και γι' αυτό η καλύτερη προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να εγγυηθεί την ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων, κάτι που είναι μια από τι θεμελιώδει ε, αξίες μας, όπως και η κυκλοφορία ε, των ανθρώπων μεταξύ συνόρων εφόσον έχουν γνήσια ταξιδιωτικά έγγραφα και μια ε, γνήσια ταυτότητα. Θα πρέπει λοιπόν τα ε, εργαλεία να εντοπίζονται ε, καταλήλως από τις αρχές εφόσον έχουν ζητηθεί σωστά και να μπορούν οι αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό θα έχει έναν θετικό αντίκτυπο. Θα προστατεύουμε τις ταυτότητες την ταυτότητα μάλλον και τα δικαιώματα των πολιτών. Πολλές φορές ε, χρησιμοποιούνται ε, πλαστά και παρανόμως οι ταυτότητες των Ευρωπαίων πολιτών ε, χωρίς να το γνωρίζουν καν. Επίση για την παρέμβαση του συναδέλφου από του Πρασίνου. Θα μπορέσουμε να βρούμε το σωστό σημείο ισορροπία μεταξύ τη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των αναγκών ασφαλεία που έχουμε. Διότι Δεν συζητάμε εδώ αλλαγέ στην μεταναστευτική μα πολιτική ή την πολιτική ασφαλεία, αλλά σημαντικέ συνιστώσει για να συνδυαστούν με άλλα εργαλεία καταπολέμηση του κλίματο. Εδώ, Πρόεδρε, απευθύνω έκκληση σε όλου σα να ενώσουμε τι προσπάθειέ μα και αύριο να υπερψηφίσουμε την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Συγγήτρια. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Το Επόμενο σημείο, δηλώσει του Συμβουλίου και τη Επιτροπή, η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικέ δραστηριότητε στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το φω των Luanda Λίξ. Σα υπενθυμίζω ότι θα έχουμε Catch the, Eye, Catch the Eye και μπλε κάρτα και με τον παραδοσιακό και με το ηλεκτρονικό σύστημα. Οδηγίε μπορείτε να βρείτε στην είσοδο του ημικυκλίου. Για τις ερωτήσεις με μπλε κάρτα σας υπενθυμίζω ότι θα επιτρέπονται μόνο αφού ακουστούν οι τοποθετήσεις των πολιτικών ομάδων. Την ε, συζήτηση θα ανοίξει η κυρία Μπρνιάτ εκ μέρους του Συμβουλίου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Σας ευχαριστώ που μας προσκαλέσατε να συμβάλλουμε σε αυτή τη συζήτηση. Να σας διασφαλίσω καταρχάς ε, να σας εγγυηθώ ότι όλα τα θεσμικά όργανα ε, επιδεικνύουν προσήλωση στην καταπολέμηση της νομοποίησης εσόδων από εγκληματικέ δραστηριότητε. Έχουμε σημειώσει πολύ μεγάλη πρόοδο μέσω και της οδηγίας για την, για την καταπολέμηση νομοποίησης εσόδων από εγκληματικέ δραστηριότητε μέσω της επικαιροποίηση του ποινικού πλαισίου. Όλα αυτοί οι νέοι κανόνες πρέπει πλέον να επιβληθούν. Οι κατηγορίες που προκύπτουν από τα Λουάντα Leaks είναι πραγματικά πολύ ανησυχητικές και θα είναι καταστροφικές αν επιβεβαιωθούν. Φαίνεται ότι ο λαός ε, μιας χώρας αλλά και επιχειρήσεις από την Ευρώπη έχουν πληγεί σοβαρότατα, έχουν ζημιωθεί οικονομικά βλέπουμε ότι οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, τόσο στην Αγγόλα όσο και στην Πορτογαλία και πρέπει να τις αφήσουμε να ολοκληρωθούν. Τον Ιούλιο η Κομισιόν κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου ε, εξέδωσε μια δημοσίευση, μια έκθεση σχετικά με παρελθοντικές περιπτώσεις ε, απάτης στον τραπεζικό τομέα. Αυτά αξιοποιήθηκαν για την επικαιροποίηση και των σχετικών κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν αποκλείεται να ξαναεμφανιστούν τέτοια φαινόμενα αν επιβεβαιωθούν οι υποψίες και οι κατηγορίες. Πέρα από τις προκλήσεις και, τις, και την επιστοδρόμηση που ενδεχομένως έχει διαπιστωθεί, υπάρχει λόγος και υπάρχει και χώρος για αισιοδοξία και για τα τρία θεσμικά όργανα διότι υπάρχει ένα κοινό επίπεδο φιλοδοξίας όσον αφορά την καταπολέμηση πλέον αυτού του φαινομένου του ξεπλήματο βρώμικου χρήματο. Τα στρατηγικά συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου το Συμβούλιο καλεί την Κομισιόν να διερευνήσει τρόπους για την ενίσχυση της εναρμόνισης των κανόνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικέ δραστηριότητε, καθώς και την αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Συμβολητικού Οργάνου. Έχουμε το σχέδιο δράσης κατά, της, ε, κατά του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος που συμφωνήθηκε στο ECOFIN το Σεπτέμβριο του 2018 και το οποίο βρίσκεται ακόμη βεβαίως σε εφαρμογή. Ταυτόχρονα η Προεδρία ξεκίνησε μια ευρύτερη ε, συζήτηση γύρω από την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της παράνομη ε, ε, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητε. Θεωρώ ότι έχουμε πλέον την ευκαιρία να κατευθυνθούμε σε ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για την καταπολέμηση των, ε, της νομιμοποίησης εσόδων και της χρηματοδότησης τρομοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό περιμένουμε τις προτάσεις Κομισιόν και ελπίζουμε ότι η Κομισιόν θα λάβει υπόψη της στο μέτρο του δυνατού και του αναγκαίου ε, όλα τα διδάγματα που προκύπτουν και από αυτή την υπόθεση των Λουάντα Λίξ. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Ντάλη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρες. Σας ευχαριστώ, Υπουργέ. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, η Κομισιόν αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η σημερινή συζήτηση και χαιρετίζει την ευκαιρία που της δίνεται να ξεκαθαρίσει την στάση της απέναντι σε ζητήματα όπως αυτά που αποκαλύφθηκαν μέσω των Λουάντα Λίξ. Συστηματικά έχουμε τονίσει ότι η καλύτερη εφαρμογή των κανόνων και την καταπολέμηση τη νομιμοποίηση όδων από εγκληματικέ δραστηριότητε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η καλύτερη εποπτεία είναι απαραίτητα στοιχεία για να ε, αυξηθεί η ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού μα συστήματο. Πέρα από τη σταθερότητα όμω, χρειάζεται να διαφυλάξουμε και την ακαιρεότητα του οικονομικού και του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος. Αυτό δεν μπορεί να είναι αρμοδιότητα ενός και μόνο κράτους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιδείξει μηδενική ένοχη στα βρώμικα χρήματα. Και θέλουμε να αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη, διάθεση, στη μας στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Επίσης, θέλουμε και να τα ενισχύσουμε τα εργαλεία αυτά. Δεν θα διστάσουμε να προτείνουμε αλλαγές στην ε, νομοθετική και ε, διοικητική δομή και αρχιτεκτονική την οποία έχουμε στη διάθεσή μας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων, της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Επίτα από το ψήφισμα του Κοινοβουλίου και τα συμπεράσματα του ΕΚΟΦΗΝ, η Κομισιόν θα εγκρίνει ένα νέο σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή των κανόνων. Πολλά έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Η πέμπτη οδηγία για την καταπολέμηση των, της νομιμοποίησης των ε, παράνομων σώδων που πρέπει να έχει μεταφερθεί στα εθνικά δίκαια έως τις 10 Ιανουαρίου δίνει καλύτερα εργαλεία ε, στα κράτη-μέλη και στην κοινωνία των πολιτών να ελέγχουν τι συμβαίνει στο πιστοτικό σύστημα, να ελέγχουν τις επιχειρηματικές συναλλαγές. Το νομικό πλαίσιο που ισχύει αποσκοπεί στο να εξασφαλίζεται η σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη να προστατεύεται η ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα και την ανάγκη να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις επιχειρηματικές χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Μέσω της δημιουργίας προσβάσιμων μητρώων, στα οποία θα καταγράφονται οι ιδιοκτήτες, η Ένωση έχει πραγματικά επιτύχει να είναι ο χρυσό κανόνα σε ολόκληρο τον κόσμο. Δυστυχώ δεν έχουν καταφέρει ακόμα όλα τα κράτη-μέλη να μεταφέρουν στο εθνικό του δίκαιο την πέμπτη ε, οδηγία για την καπτολέμηση τη παράνο... της νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Σήμερα η Κομισιόν ξεκίνησε διαδικασία επιπαραβάση κατά 8 κρατών που δεν το έχουν πράξει ακόμα. Όμω το πρόβλημα δεν είναι τόσο η έλλειψη των κανόνων. Είναι η επιβολή, η εφαρμογή αυτών των κανόνων. Και το γεγονό ότι η εφαρμογή αυτή γίνεται σε επίπεδο εθνικό και γίνεται με ανομοιόμορφο τρόπο. Οι πρόσφατες αλλαγές στο πλαίσιο που διέπουν τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές δίνει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να καθοδηγεί τους, τις εποπτικές αρχές της Ευρώπης όσον αφορά τον εντοπισμό της, των περιπτώσεων ε, ε, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικέ δραστηριότητε. Η Κομισιόν βεβαίω αναγνωρίζει ότι πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα. Χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε διαρθρωτικέ αδυναμίε που σχετίζονται με τον διοικητικό κατακαιρματισμό μεταξύ των κρατών μελών. Εδώ ακριβώ υπάρχει και η ευρωπαϊκή προστιθόμενη αξία. Η Κομισιόν επιδιώκει να εργαστεί προς την οικοδόμηση ενός ενιαίου ολοκληρωμένου συστήματος καταπολέμησης της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και να επιφέρει σε αυτό το σύστημα όλες τις απαραίτητες ε, βελτιώσεις. Υπάρχει περιθώριο εναρμόνισης των υφιστάμενων κανόνων. Χρειάζεται καλύτερη ανταλλαγή από ε, πληροφοριών μεταξύ των διοκτικών αρχών, ώστε να εντοπίζονται και να συλλαμβάνονται οι εγκληματίες και για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων. Ε, ε, ένα τέτοιο επικαιροποιημένο σύνολο νέων κανόνων θα δώσει μεγαλύτερο ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την εποπτεία όλων αυτών των δραστηριοτήτων. Και αυτό είναι τελειωμένο, γιατί αυτό αφορά και τον, την εποπτεία και τον συντονισμό των ε, οικονομικών ε, αστυνομικών αρχών. Είναι λοιπόν απαραίτητο να δημιουργηθεί μια τέτοια δομή. Όμως η δημιουργία μιας δομής δεν πρέπει να είναι αυτός σκοπός ο φορέα, είτε θα είναι καινούριο, είτε θα βασίζεται μέσω της διεύρυνση αρμοδιοτήτων ή φυστάμενου φορέα, θα πρέπει να έχει συγκεκριμένο πεδίο ισχύω, αρμοδιότητες και αποτελεσματική διακυβέρνηση. Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να βασιζόμαστε στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να καταλήξουμε σε ένα πιο αποτελεσματικό σε μια πιο αποτελεσματική αρχιτεκτονική όσον αφορά την εποπτεία. Αυτή είναι και η φιλοδοξία μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Εκ μέρους των πολιτικών ομάδων τώρα, εκ μέρους του ΕΛΚ, ο κύριος Φέρμπερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, Επίτροπε, που είστε εδώ. Η υπόθεση Λουάντα Λίξ δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με πέντε ε, οδηγίες ε, για, την, για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος τελικά καταφέρνει το φαινόμενο αυτό να μην το καταπολεμεί ε, και παραμένει ελκυστικό. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα γιατί Κύριε Επίτροπε, συμφωνώ ότι είναι μεγάλο το κέρδος από το ξέπλυσμα του βρώμικου χρήματος. Θα πρέπει να ε, δούμε την τελευταία φορά στις 10 Ιανουαρίου. Πέντε από τα 25 χρόνια έχουν υλοποιήσει και μεταφέρει πλήρως την ε, οδηγία. Και ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ενημερώσει καν για την μεταφορά και την υλοποίηση. Επιτέλου, θα πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία για τα κράτη αυτά. Όμω το θέμα είναι πώ στην πράξη εφαρμόζουν ω επιβάλλει οδηγία και τι κάνουν για το ξέπλυμα το βρώμικο χρήματο. Ε, έχουμε πολλά ωραία ψηφίσματα ε, και αποφάσει των ε, Υπουργών Οικονομικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά προφανώ τα κράτη-μέλη δεν είναι ακόμα σε θέση να καταπολεμήσουν δραστικά το φαινόμενο αυτό. Και θα πρέπει επιτέλους να σκεφτούμε πώς μπορεί να βρεθεί μια λύση και να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, που πάλι φορέσατε τα ακουστικά σα και με ακούτε. Ε, και τώρα ε, το θέμα είναι η ακαιρεότητα του ευρωπαϊκού οικονομικού συστήματος, η ασφάλεια των πολιτών μας, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο, τα οποία όλα είναι αλληλένδετα. Απευθεία αλληλένδετα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ε, πώς μπορούμε τα αξιόπινα να τα καταπολεμήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τη δημιουργία μια κατάλληλη αρχή. Θα πρέπει, αρχής, θα, πρέπει τα ευρωπαϊκά κράτη να συνεργαστούν για να βρεθεί μια ε, κοινή αντίληψη του φαινομένου αυτού και ένα συντονισμός για την καταπολέμηση. Ε, ευχαριστώ. Εκ μέρου ε, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο κύριο Χέινα Λουόμα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για άλλη μια φορά θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τους δημοσιογράφους, τους ανεξάρτητους δημοσιογράφους, οι οποίοι προέβησαν σε αυτές τις ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες για αυτή την ε, φυγή κεφαλαίων. Βλέπουμε λοιπόν ότι πρέπει να στραφούμε προς τα εκεί. Μιλούμε για δύο δολάρια την ημέρα που διαφεύγουν και μιλούμε για εκατοντάδες εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων που ε, φεύγουν. Ε, και ένα σωρό νομικοί έχουν ανακατευτεί για να βοηθήσουν σε αυτό το σκάνδαλο ακόμα και δημόσια υπάλληλοι. Οπότε εμείς αυτό που θέλουμε είναι να αλλάξουν οι κανόνες του παιχνιδιού. Θα πρέπει να γίνουμε πολύ αυστηρότεροι. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπουμε τέτοια πράγματα. Εντάξει με την οδηγία, αλλά χρειάζεται νομοθεσία κοινή και θα πρέπει ο τραπεζικός κόσμος επίσης να ε, συμμορφωθεί. Καλύτερη υποπτία πανευρωπαϊκά. Ο πρόεδρος για το Renew Europe. Η κυρία Στρουγκάριο για δύο λεπτά. Δεν έχετε ανάψει το μικρόφωνο. Ευχαριστώ, θα σας τα πω ρουμανικά. Δεν γίνεται πλήρως και σωστά η μεταφορά στο ιστορικό δίκαιο των οδηγιών για να καταπολεμηθεί ε, το ξέπλυμα χρήματος. Σήμερα ε, ξεκίνησε η διαδικασία επί παραβάση κατά διαφόρων χωρών και κατά της Ρουμανίας γιατί δεν είχε γίνει σωστά η μεταφορά της πέμπτης οδηγίας. Αλλά πολλά κρατήματα... μέλη ε, δεν μετέφεραν την τέταρτη ομιλία που είχε, οδηγία που είχε προθεσμία το 2017 και τώρα ξυπνήσαμε με το σκάνδαλο Λουάντα Λίξ. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τη διάθεση προϊόντων εγκλήματος, ε, χρειάζεται θάρρος, είναι κάτι που επιβάλλεται, αλλά δεν αρκούν οι οδηγίες. Θα πρέπει να αλλάξει κατάσταση πραγμάτων και να δούμε ποιοι είναι οι τελικοί ε, ωφελούμενοι από όλη αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν κάποια κενά στην νομοθεσία που μας κάνουν ε, τους Ένωση και κρατημέλη. Είναι απαράδεκτο μια μεγάλη εταιρεία παροχής συμβουλών που εργάζεται και για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να δουλεύει για λογαριασμό δικτατόρων αυτών των τρίτων χωρών και να τους βοηθά να μεταφέρουν τα χρήματά τους σε φορολογικούς παραδείσους και να φοροδιαφεύγουν. Χρειάζεται επομένω μια στιβαρή στεγανή νομοθεσία, ε, ακριβώς όπως τα είπαμε τον ε, Δεκέμβριο. Και η ερευνητική δημοσιογραφία για άλλη μια φορά απέδειξε πόσο σημαντικό είναι το έργο της όσον αφορά το ξέπλυμα. Ε, άρα θα πρέπει να το έχουμε το θέμα αυτό ως προτεραιότητα και στο νομοθετικό έργο μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εκ μέρους των Πρασίνων ο κύριος Γκίγκολτ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Παρακολουθώντας την δημόσια συζήτηση μετά τις αποκαλύψεις Λουάντα Λίξ, πραγματικά δημιουργούνται αρνητικά συναισθήματα. Μου φαίνεται ότι ε, έχουμε αρχίσει και συνηθίζουμε τέτοια φορολογικά σκάνδαλα. Δεν υπάρχει ίδια αναταραχή, ε, φαίνεται ότι οι πολιτικοί δεν έχουν τελικά καμία εξουσία απέναντι σε μια τεράστια βιομηχανία φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής για κάποιους λίγους πλούσιους. Όμως οι πολιτικοί δεν πρέπει ποτέ να σταματήσουμε να καταπολεμούμε την αδικία. Ούτε να φοβόμαστε να πληγεί η δημοκρατία μας, όσο ισχυρή και πλούσιοι κι αν είναι οι αντίπαλοι. Γιατί και σε αυτή την περίπτωση δεν είναι τυχαίο και στα Λουάντα Leaks ότι η Πορτογαλία και με τα Football Leaks πριν από ένα χρόνο η Πορτογαλία βρέθηκε στο επίκεντρο ε, των κατηγοριών. Τι έγινε τελικά, ο πληροφοριοδότης βρέθηκε στη φυλακή και οι ε, αδικοπραγούντες τελικά έχουν ξεφύγει. Χιλιάδες ε, ε, είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν καταφύγει στην Μαδέρα με, τις, με τα περιουσιακά του στοιχεία. Αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να επιβάλλει το ευρωπαϊκό δίκαιο σε όλα τα κράτη-μέλη και δεν μπορεί να περιμένει με την έναρξη διαδικασιών επί παραβάση. Δυστυχώς παρακολουθούσα άπραγη τα όσα συνέβαιναν στην Πορτογαλία ενώ εξελίσσονταν τεράστια σκάνδυλα, δεν καταδικάζονταν οι ε, εγκληματίες. Έχουμε πρόβλημα κράτους δικαίου στην Πορτογαλία και πρέπει η Κομισιόν γρήγορα με στοχευμένες διαδικασίες επιπαραβάση να το αντιμετωπίσει. Και η, χρειαζόμαστε επίσης μια νέα οδηγία για τους οικονομικούς ελεγκτές, ώστε οι οικονομικοί ελεγκτές πλέον να μην μπορούν να εμπλέκονται σε τέτοιου είδους οικονομικά σκάνδαλα όπως αυτά που αποκαλύφθηκαν στα Λουάντα Leaks. Το πρόβλημα δεν έχει λυθεί, πρέπει να συνεχίσουμε να το καταπολεμούμε. Ευχαριστούμε. Εκ μέρους του ECR, η κυρία Κέμπα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Μόνο σκληρή νομοθεσία που θα προβλέπει συγκεκριμένε κυρώσει μπορεί να μα οδηγήσει στην πρόληψη του οργανωμένου εγκλήματο. Στην Πολωνία έχουμε θεσπίσει σχετικούς κανόνες υπό τον Σπίγνιος Μπράζδο, τον Γενικό Εισαγγελέα και έχουμε καταπολεμήσει αποτελεσματικά την ε, νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Αυστηρήναμε το νομοθετικό πλαίσιο και καταφέραμε να ανακτήσουμε ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Πρόκειται για ζήτημα του πόσο προσιλωμένε είναι οι εισαγγελικέ αρχές και τα Υπουργεία Δικαιοσύνη. Εμείς στη χώρα μου έχουμε πλέον μια σειρά από εργαλεία στη διάθεσή μας, κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, πάγωμα τραπεζικών λογαριασμών, υπερορισμοί περιορισμοί σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δεν συνεργάζονται. Έχουμε μια σειρά από στοιχεία, μηχανισμού, εργαλεία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο και του ξεπλήματο βρώμικου χρήματο στην Πολωνία. Φυσικά, η πέμπτη οδηγία για την καταπολέμηση τη ε, νομοποίηση παρανόμων εσόδων είναι ένα ευρωπαϊκό εργαλείο εξαιρετικά σημαντικό που μπορεί επίση να χρησιμοποιηθεί στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο. Ευχαριστώ πολύ. Μέρο τη ΚΟΕ, ο Για ένα μισό λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το σκάνδαλο του Λουάντα Λίξ προκαλώ προφανώς ε, έχει να κάνει με πολλές εθνικές ευθύνες και στη χώρα μου επί πολλά χρόνια η ελίτ της οικονομίας και της πολιτικής δεν αισθάνονταν κανένα πρόβλημα λόγω των εμπορικών κινήσεων της Ιζαμπέλ του Σάντους. Οι ε, εθνικές δικαιοδοσίες, η δικιά μας, η Μάλτα, συνεργάστηκαν για όλο τον κύκλο αυτοξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Ε, εδώ υπάρχουν ευθύνε και από την πλευρά των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων όμω. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αν υπάρχουν εθνικέ δικαιοδοσίε που διευκολύνουν την λεύκανση παράνομων εσόδων, την φοροδιαφυγή, το οργανωμένο οικονομικό έγκλημα, τότε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικώ το σύνολό της Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει γνώση και να το καταπολεμήσει. Ο κίνδυνος από τα σκάνδαλα αυτά που καταλήγουν στην ατιμορρησία και χωρίς συνέπειες για όσους ε, ήταν δράστες στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος είναι κάτι που δεν πρέπει να ε, επιτρέπεται. Οι όμιλοι χρηματοπιστωτικοί, αυτοί που ε, πολλές φορές ε, προσλαμβάνει με σύμβαση η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναλάβουν υπηρεσίες της. Αυτά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένοχοι. Αν τίποτε από αυτά δεν έχει συνέπειε, εάν στο τέλο αυτή τη διαδικασία ο μόνο που θα κατηγορηθεί είναι ο, ο κατηγορούμενος ή αυτός που ήταν ο καταγγέλων και δημοσιοποίησε τα σχετικά έγγραφα, τότε αυτό που φαίνεται είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει ατιμορρησία σε όσους έχουν διαπράξει αξιόπινες πράξεις. Ευχαριστούμε. Εδώ κλείνει ο κατάλογος των αγορητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Επόμενη κυρία Περέιρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ε, το λεύκανση παράνομων προσώπων είναι ένα πολύπτυχο ε, έγκλημα γιατί έχει να κάνει με περιουσιακά στοιχεία και την συμμετοχή εταιριών καθώς και τη στρέβλωση του οικονομικού κύκλου. Ε, το βρώμικο χρήμα δεν χάνει ποτέ την καταγωγή του που είναι ε, αξιόπινη εγκληματική. Θα πρέπει λοιπόν να ε, δούμε όχι απλώς τα θέματα εποπτείας ή νομικών διαθετήσεων, αλλά ότι είναι θέμα κράτους δικαίου να το καταπολεμήσουμε το φαινόμενο αυτό με αποφασιστικές και δραστικές κινήσεις. Θα πρέπει η πέμπτη οδηγία για την καταπολέμηση του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος να μεταφερθεί σωστά. Λείπει η αποφασιστικότητα λείπει η τόλμη από τα 27 κράτη-μέλη, όπως είπε και η Επίτροπο στην αρχική της παρέμβαση. Ε, η πόρτα παραμένει μισά ανοιχτή για να περάσουν ε, οι θράστες. Το Κοινοβούλιο λοιπόν θα πρέπει με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα να αντιδράσει και θα πρέπει να μην περνάνε οδηγίε και κανονισμοί σμάτιν αλλά να ενισχύσουμε το Ευρωπαϊκό Κεντρικό Σύστημα και ε, όχι να αφήνουμε τους εθνικούς ε, μεταρρυθμιστές ε, στην τύχη τους ή να αποτυγχάνουν. Ευχαριστούμε κυρία Κινίτση για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι αποκαλύψεις του Λουάντα Λίξ εμπλέκουν και κάποιους από τα κράτη-μέλη. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε έχουμε προτεραιότητα την κατολέμηση του ξεπλήματος ε, σχετίζεται με απάτη και είναι ένα μέσο ούτως ώστε και οι οργανώσεις, οι εγκληματικές να υποσκάπτουν την οικονομία και τον ανταγωνισμό. Είναι τρόπος επίσης χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, οπότε θα πρέπει να θωρακίσουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά του ξεπλήματος και να εναρμονιστούν οι σχετικές εθνικές νομοθεσίες ε, και να εφαρμοστούν οι οδηγίες για αυτό το θέμα και στο ποινικό δίκαιο. Θα πρέπει ε, επίσης ε, η έρευνα να μπορεί να έχει πρόσβαση παντού και θα πρέπει οι διοικητικές αρχές να μπορούν να κάνουν έλεγχο και σε διοικητικό επίπεδο. Ε, αυτό το οποίο κάνουμε στην Ιταλία με την οικονομική μας αστυνομία Guardia di Finanza και να δούμε τι γίνεται με τα προϊόντα εγκλήματος, τα οποία όπως γνωρίζουμε τώρα ότι ανέρχονται στο 1% της οικονομίας. Ευχαριστούμε κυρία Κινίτση, λέει ο Πρόεδρος, αγαπητή Κατερίνα. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Γκερέιρου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το σκάνδαλο Λουάντα Λίξ δείχνει πως ε, το χρηματοπιστωτικό ε, σύστημα αφήνει παραθυράκια για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και την ε, παρανομία. Ε, αυτό το σύστημα λειτουργεί εδώ και 7 χρόνια στην Πορτογαλία, επιτρέποντας να πέσουν θύματα η πλειοψηφία των πολιτών. Το χρηματοπιστωτικό αυτό σύστημα που καταργεί ε, θέσεις εργασίας και εμπλέκει 17 εταιρείε τουλάχιστον στην περίπτωση αυτή το Ευρωκοινοβούλιο με τις θεωρήσεις που έχουν μοιραστεί σε όλο τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά σοβαρά υπόψη όμω το Λουάντα Λίξ δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με αδιαφορία από το πολιτικό σύστημα. Πρέπει να υπάρξει άμεση μεταφορά τη πέμπτη οδηγία για το πιο πλευρόμικο χρήματο, ιδίω στην Πορτογαλία, να προστατεύονται οι καταγγέλλοντε και όλη η ερευνητική δημοσιογραφία να προστατεύεται στι χώρε, γιατί αυτοί είναι θεματοφύλακε τη δημοκρατία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, συνάδελφο. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριο Φεραίρα. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα, χρηματικά, τα οικονομικά σκανδαλά όπως το Λουάντε Λίξ δείχνουν ότι υπάρχει αδιαφάνεια, ανωνυμία και ακόμα διακίνηση μεγάλων κεφαλαίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θύμα και όμοιρο των ε, οικονομικών συμφερόντων των πολυεθνικών και όχι μόνο. Θα πρέπει να, πάρουμε αποφα... Ε, να κάνουμε αποφασιστικέ κινήσει για την καταπολέμηση του ξεπλήματο βρώμικου χρήματο. Παρ' όλα αυτά, για την ώρα δεν έχει αλλάξει τίποτα. Θα πρέπει λοιπόν οι αρχές των ε, κρατών μελών να κοιτάξουν πώς λειτουργούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και αν ε, λειτουργούν νόμιμα. Δεν επιτρέπονται τέτοιες ε, κινήσεις, ούτε υποκριτικές κινήσεις παρεμβατισμού που τρέπουν σε ευρωπαϊκές δυνάμεις να ικανοποιήσουν τις νεοαπικροκρατικές τους ε, ορέξεις. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να λυθεί ο κόμβος που, θα πρέπει, ε, που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ των φορολογικών ε, σχέσεων που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποιες χώρες, όπου έχουν δημιουργηθεί ιδιαίτερες προνομιακές σχέσεις. Αυτός ο κόμμος πρέπει να λυθεί. Ευχαριστούμε συνάδελφε Φερέρα και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Ράντεφ. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε αυστηρούς κανόνες. Αυτούς κανόνες κατά πολέμησης ε, του ξεπλήματος χρήματος και όσον αφορά επίσης λαθροχειρίες στο τραπεζικό σύστημα και αυτά τα συζητήσαμε και τον Ιανουάριο φέτος, αλλά το σκάνδαλο αυτό που ξέσπασε σημαίνει ότι οι σχετικοί κανόνες δεν έχουν ακόμα υιοθετηθεί από τράπεζες και από κάποια κρατημέλη. Επομένως, χρειάζεται να ε, υπάρχει αυστηρή νομοθεσία και να έχουμε τα απαραίτητα μέσα, ούτω ώστε να καταστήλουμε κάθε ύποπτη δραστηριότητα. Ε, ε, αλλιώς όλες οι προσπάθειές μας πέφτουν στο κενό. Δεν είναι μόνο η απειλή απ' έξω. Έχουμε ξέβλημα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε η χρηματοοικονομική μας αγορά πέφτει θύμα αυτών των εγκληματιών. Το Ρόντε είναι ένα παράδειγμα του τι γίνεται όταν δεν εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο. Είναι θέμα και ελέγχου τη ταυτότητας των πελατών, των τραπεζών, είναι θέμα καταγγελίας ε, και αναφοράς υπόπτων συναλλαγών κλπ. Άρα χρειάζεται να τηρήσουμε την νομοθεσία και να υπάρξει έλεγχος του αν εφαρμόζεται. Ευχαριστούμε στην αδελφή ο Πρόεδρος. Και τώρα, ο κύριος Μάρκης, έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, με αυτή την τόσο επίκαιρη συζήτηση ξαναβλέπουμε ένα από τα βασικά προβλήματα αυτού του Κοινοβουλίου. Οι πρακτικές αυτές πλήττουν την ευρωπαϊκή κοινωνία, διότι ακριβώς σημαντικά τμήματα των ε, κεφαλαίων μας ε, προέρχονται από, ε, μάλλον πηγαίνουν σε παράνομε ενέργειε, σε ψηφιακέ συναλλαγέ, γενικώ οι συναλλαγέ κάθε μέρα γίνονται και πιο αδιαφανεί και ε, με εξελιγμένα ε, τεχνολογικά μέσα οι τρόποι παρακολούθηση και ελέγχου που έχουμε ως τώρα δεν ήταν αποτελεσματικέ. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα νέο ορισμό των παράνομων συνελεγών και χρηματοπιστωτικών κινήσεων και να έχουμε καλύτερη συνεργασία μεταξύ των αρχών των 100 μελών. Θα πρέπει να ενισχύσουμε το ρόλο των ευρωπαϊκών αρχών και θα πρέπει η συμμόρφωση με του κανόνε να ισχύει καθώ και, ε, και για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και για τι διεκτικέ αρχέ των 100 μελών. Θα πρέπει λοιπόν να επιταχυνθεί η ρυθμιστική και νομοθετική διαδικασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο επίπεδο και σύντομα να εγκριθεί ένα ευρωπαϊκό κανονισμό και εν τέλει θα πρέπει ο κόσμο να μπορεί να εμπιστεύεται το τράπεζε και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τι ε, κρατικέ αρχέ. Ε, να συνεχίσουμε αυτόν τον ε, αξιέπαινο αγώνα. Ευχαριστούμε συνάδελφε Μάρκες και τώρα ο κύριος Κάζα. Παρακαλώ κύριε Κοσμή τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το ξεκινάμε χρήματο παραμένει ένα έγκλημα που θα πρέπει να καταπολεμηθεί, αλλά είναι δύσκολο ναι, να επισημανθεί ακριβώ ε, ποιοι θα πρέπει να διωχθούν για αυτές τις εγκληματικέ δραστηριότητε. Ε, χρειάζονται κάποια στοιχεία που να έχει η, η εισαγγελία και να μην ε, οδηγούμαστε σε ατιμορρησία των ενόχων και η Δάφνη Καρβάνα ήταν ε, ερευνητική, στην ερευνητική δημοσιογραφία και προσπαθούσε και αυτή κάτι να, τέτοιο να καταφέρει. Ε, όμως το θέμα είναι ότι δεν υπήρχαν όλα τα στοιχεία και επομένω δεν μπορούσαμε να αποδώσουμε δικαιοσύνη και θα πρέπει τα σχετικά στοιχεία να πηγαίνουν όπου χρειάζεται. Ε, μεταξύ των διοικητικών αρχών, ούτως ώστε να υπάρχει συνεργασία και με τις τρίτες χώρες όσον αφορά το ξύλινο του χρήματος. Θα πρέπει επίσης να επιβαλούνται ποινές για όποιον δεν συνεργάζεται με την δικαιοσύνη και τις διοικητικές αρχές, να μην συνεχιστεί και η τρέχουσα κατάσταση. Ευχαριστούμε, αγαπητέ συνάδελφε. Και τώρα ο κύριος Τάγκ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο ήταν αυτά τα οποία έκλεψε από τον λαό της Αγγόλας ε, ε, αυτή. Και η ε, Ισαβέλ Σάντος έγινε μία από τις ε, πλουσιότερες γυναίκες και αυτό μέσω της διαφθοράς, ότι αυτό φταίει. Αλλά όμως αυτό το οποίο έκανε ήταν να πάρει αυτά τα λεφτά για να τα ξοδέψει εδώ. Ήταν Ολλανδικό το γιο του που είχε των 50 εκατομμυρίων. Ε, και είχε επίσης επενδύσει στο Λονδίνο Επομένως, αυτοί που πήραν τα λεφτά είναι οι εγκληματίες. Οι τραπεζίτες του Λουξεμβούργου, του Λίχτενστάιν, εταιρείε από το Άμστερνταμ, ε, την πόλη μου, γιατί ε, κυκλοφορούν ελεύθεροι όλοι αυτοί οι εγκληματίες. Ο Πίντο, ε, αυτός που έβγαλε στη φόρα αυτά τα σκάνδαλα, είναι στη φυλακή επί ένα χρόνο. Είναι ένας καταγγέλων που αξίζει προστασίας. Αυτά συγκεκριμένα θέλω να απευθύνω σε ερωτήμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι δικό μας. Θα πρέπει να προστατεύσουμε εκείνους οι οποίοι βγάζουν στη φόρα αυτά τα εγκλήματα. Να καταπολεμήσουμε το ξέβλημα, να προστατεύσουμε τις ε, πηγές μας, να δώσουμε την ε, μάχη. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφε. Και τώρα, το λόγο έχει ο Αντιπρόεδρος Κάρας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Αντιπρόεδρε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι. Δύο-τρεις δολάρια ξεπλένονται κάθε χρόνο στον κόσμο. Όμως δεν αρκεί να κοιτάμε μόνο έξω από το σπίτι μας. Το πρόβλημα υπάρχει και εδώ. Πάνω από 110 δισεκατομμύρια ευρώ ξεπλένονται ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποσό σχεδόν εισάξιο με τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Άρα πρόκειται για ένα ζήτημα που σχετίζεται και με την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας. Είναι πραγματικά ανατριχιαστικό το γεγονός ότι υπάρχει ακόμη ε, μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις υποχρεώσεις των κρατών μελών και τα όσα τελικά κάνουν. Είναι απαράδεκτο το γεγονό ότι υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν μεταφέρει ακόμα στο εθνικό του δίκαιο την τέταρτη οδηγία, ενώ έχουμε ήδη θεσπίσει την πέμπτη οδηγία. Ότι ακόμη χρειαζόμαστε ε, μια εποπτεία ε, για την καταπολέμηση τους, ε, της, ε, του ξεπλήματος χρήματος. Ότι χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή οικονομική αστυνομία. Τα έχουμε υποσχεθεί αυτά εδώ και πολλά χρόνια. Ας τα κάνουμε επιτέλους. Ευχαριστώ πολύ. λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά τις ε, συζητήσεις που έγιναν για τα Panama Papers, τα Paradise Papers, τα Lux Leaks και όλα αυτά τα σκάνδαλα, να που για άλλη μια φορά βρισκόμαστε εδώ να συζητούμε αυτή τη φορά τα Luanda Leaks. Δεν έχει νόημα να συζητήσουμε τι λεπτομέρειε τη υπόθεση τη κυρία Ντο Αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι να εξετάσουμε τα, τα του οίκου μα. Το Ντουμπάι πολλές φορές αναφέρονται, αναφέρεται ως προορισμός για ξέπλυμα ε, βρώμικου χρήματος. Γιατί λοιπόν τα Εμμυράτα δεν βρίσκονται στο μαύρο κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ καλώ την Κομισιόν να το εξετάσει αυτό το ζήτημα όταν θα αναθεωρήσει τους καταλόγους αυτούς. Δεύτερον, σε πορτογαλική τράπεζα και Μαλτέζη χρηματοπιστωτική φορείς βοήθησαν την κυρία Σάντος να αξιοποιήσει διάφορα παραθυράκια και να ξεπλύνει χρήμα. Τα νομοθετικά, ε, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να κατευθυνθούν και σε αυτά. Μπορούμε να κάνουμε κριτική βεβαίως στην πλουσιότερη γυναίκα της Αφρικής, όμως πρέπει να αναρωτηθούμε και εδώ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί επιτρέπουμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε συνάδελφε και τώρα ξεκινώ τη δικασία Κατστιάη. Έχω δεχτεί πέντε αιτήματα, και θα τις αποδεκτώ όλες. Ξεκινάμε με την κυρία Πίτι Κάινεν για ένα λεπτό. Παρακαλώ. Γνωρίζουμε όλοι ότι η μεγαλύτερη ευθύνη για την εφαρμογή των οδογιών αυτών ε, εναπόκειται στα κράτη-μέλη. Και αυτό ε, στερεί την Ευρωπαϊκή Ένωση από αρμοδιότητες όσον αφορά τον συντονισμό μεταξύ των ε, ευρωπαϊκών ε, οικονομικών αστυνομιών. Πρέπει επιτέλους να θεσπιστούν νέα πρότυπα. Το σύστημα δεν λειτουργεί ακριβώς γιατί έτσι έχει σχεδιαστεί. Αυτός είναι ο λόγος που για άλλη μια φορά διαπιστώνουμε πόσο αναποτελεσματικοί είμαστε. Ελπίζω λοιπόν ότι η Κομισιόν σοβαρά θα εξετάσει ε, το ενδεχόμενο να τροποποιήσει την οδηγία για την καταπολέμηση του ξεπλήματος ε, χρήματος και να την μετατρέψει σε κανονισμό με τον οποίο θα ενισχυθεί η διαφάνεια των μητρών ιδιοκτητών, θα ενισχύσει την Ευρωπαϊκή επίπεδο για να υπάρξει ένα πραγματικά λειτουργικό σύστημα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε συνάδελφε και τώρα ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ για ένα λεπτό πάλι. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε τελείω καλώ ορίσατε σε αυτή τη ε, συζήτηση κατά τη διάθεση προϊόντο εγκλήματο. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε. Υπάρχει προστορία γιατί πριν το Λόντε το Λουξ Λίξ και τα Πάναμα Λίξ Είχαμε μια ερευνητική επιτροπή εδώ πέρα. Εγώ δούλευα εκεί και καταλήξαμε σε κάποιες προτάσεις προς την Κομισιόν με κάποια συμπεράσματα. Οπότε από την τέταρτη οδηγία φτάσαμε στην πέμπτη οδηγία και έτσι έχουμε περισσότερη διαφάνεια και έχουμε περισσότερο εντοπισμό των ε, δικαιούχων λογαριασμών. Γιατί όλα αυτά τα οποία αναφέρονται ε, συνεχώς χειροτερεύουν ε, την κατάσταση αυτή όσον αφορά την ε, διαφθορά, όσον αφορά την ε, απάτη, το ξέβλημα. Αυτό είναι χειρότερο ότι έχουμε τώρα την κόρη του Πρόεδρου, την πιο πλούσια γυναίκα της Αφρικής. Και θα πρέπει να προστατεύονται οι καταγγέλλοντες γιατί είναι αφόρητο αυτό το να μην έχει γίνει η μεταφορά στην Πορτογαλία της οδηγίας και ο Ρούι Πίντο, ο οποίος έκανε την αποκάλυψη, τώρα βρίσκεται φυλακισμένος ε, δεν θα πρέπει αυτός να είναι στη φυλακή. Θα πρέπει να είναι εγκληματίε στη φυλακή. Ο Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ κύριε συνάδελφε. Και τώρα τον λόγο έχει ο κύριος Μπρουσίνσκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είπαμε μία σειρά πράγματα απόψε γιατί για άλλη μια φορά συζητούμε τα σκάνδαλα και θα πρέπει να αναλογιστούμε το ότι το ξέπλυμα δεν μόνο στον τρίτο κόσμο, δεν μόνο στην Αφρική και στους φορολογικούς παραδείσους, διότι παραδόξως ε, αυτοί που ωφελούνται από αυτή την κατάσταση επενδύουν και ξοδεύουν τα χρήματα αυτά στην Ευρώπη. Και ούτε δικαιωτικές αρχές, ε, ούτε δικαιοσύνη στις χώρες μέλη δεν μπορούσαν κάτι να κάνουν. Είχαμε έξι χώρες που συνεννοήθηκαν πέρσι και έφτιαξαν μια υπηρεσία για το ξύλωμα του χρήματος και εγώ μπορώ να σας πω μια που έχω διατελέσει υπουργό Εσωτερικών στην Πολωνία ότι η επιτυχία ε, των υπηρεσιών αυτών οφειλόταν στην συνεργασία με άλλες χώρες και με ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Μόνο αυτό είναι η λύση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ συνάδελφα. Και τώρα. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η νομοθεσία κατά του ξεπλήματο βρώμικου χρήματο από τα κάτι μέλη θα πρέπει να γίνει αυστηρότερη. Ε, πρέπει να περιοριστεί ο χώρο για τα καζίνο και τα παίγνια. Όμω, βλέπουμε ε, το οργανωμένο οικονομικό έγκλημα να δρά τα πλοκάμια του διεθνώς και να έχουν δυσκολίες τα κατημέλη να το ελέγξουν. Η ερώτησή μου είναι εάν υπάρχουν περιττέρω ιδέες για να πατάξουμε αυτό το είδους την εγκληματικότητα και το ξέπλυμα χρήμα. χρήματο. Ευχαριστώ. Και ε, τελευταία στιγμή έχω λάβει κι άλλο ένα αίτημα από τον κύριο Μάντελς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όλο και περισσότερο το ξέβλημα βρώμικου χρήματο ε, είναι κάτι που το αναλαμβάνουν μεγάλε τράπεζε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υπάρχουν ακυρώσει, ε, δεν υπάρχουν ποινέ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε συνάδελφε. Λίγη η συζήτηση και όπως προβλέπετε για να απαντήσει δίνουμε το λόγο. Α, όχι, ξέχασα. Με συγχωρείτε. Έχω και ένα αίτημα από τον κύριο Πόλτσακ. Παρακαλώ κύριε Πόλτσακ. Το πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, εδώ μιλάμε για διεθνείς εγκληματικές δραστηριότητες και δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε. θα πρέπει να προστατεύσουμε τους καταγγέλλοντες και τους ερευνητές δημοσιογράφους διότι η διεθνή τους, η διεθνής τους προστασία είναι ένα πρόβλημα. Βεβαίως, ευρωπαϊκές τράπεζες ε, και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν αποκρύψει τέτοιες παράνομες δραστηριότητες για τα παράνομα έσοδα από την Αγγόλα. Έχουμε πέντε σχετικές οδηγίες. Θα πρέπει να κοιτάξουμε την καλύτερη και ομοιογενέστερη ε, μεταφορά τους για να υπάρχουν ε, οι κατάλληλες δυνατότητες αντίδρασης, οι κατάλληλες αρμοδιότητες. Θα πρέπει, όχι απλώς να τα λέμε εδώ, να γίνει ότι πρέπει και στο τομέα που χρειάζεται. Ευχαριστούμε κύριε Πόλτσακ. Και επιτέλους μπορώ να κηρύξω τη λήξη της συζήτησης και να δώσω το λόγο στην Επίτροπο Ντάλη για την απάντησή της. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το γεγονό ότι αφιέρωσε χρόνο να γίνει αυτή η συζήτηση για αυτό το πολύ επίκαιρο θέμα, καθώ και για την αφοσίωσή του στην ενίσχυση, περαιτέρω ενίσχυση όλων των εργαλείων μας που έχουμε για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Πρέπει να δράσουμε επί όλων αυτών των πορισμάτων, ευρημάτων και νομίζω ότι μπορούμε να ε, περιγράψουμε ήδη ε, τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα της Ένωσης. Και είμαστε αποφασισμένοι να συνεργαστούμε με διεθνείς εταίρους και σε καινοτόμε λύσεις. Και είναι πραγματικά κρίσιμη σημασία να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο να εφαρμόζεται πλήρω και ορθώς. Και σε αυτό βεβαίως συμπεριλαμβάνεται και η προστασία των πληροφοριοδοτών. Να δοθούν νέα κίνητρα στον ρόλο της Ένωσης όσον αφορά τον συντονισμό και την αποτελεσματική δράση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε, ε, σας ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε. Και τώρα ο λόγος στην κυρία Μπρνιάκ. Ευχαριστώ αξιότιμοι ευρωβουλευτέ. Παρακολούθησα τη συζήτηση με μεγάλη προσοχή και άκουσα και την τοποθέτηση της Κομισιόν. Δράτω με αυτή τη ευκαιρία για να επιβεβαιώσω την σημασία που δίνει η Προεδρία στην καταπολέμηση τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων και τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία και προσβλέπω στη συνεχιζόμενη συνεργασία μα. Η Προεδρία θα είναι πάντοτε στη διάθεσή σα σε οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση που γίνει στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. discussione è chiusa. Ευχαριστούμε κύριε Πορχέ, Λίγη συζήτηση. Συνάδελφοι, έχω μερικές ανακοινώσεις να σας κάνω. Ο κύριος Ντάντι άφησε την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και θα προσχωρήσει στην ομάδα Renew. Από τις 13 Φεβρουαρίου 2020 θα ισχύσει αυτό. Δεύτερη ανακοίνωση, συνάδελφοι, σας παρακαλώ. Συνάδελφοι, παρακαλώ. Κύριε Γκίγκολντ, κύριε Κάρα, παρακαλώ ησυχάστε. Η ομάδα Renew Europe ενημερώνει το Προεδρείο για κάποιε τι αποφάσει που αλλάζουν τη σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπιών. Οι αποφάσει αυτέ θα ισχύουν από 13 Φεβρουαρίου 2020. Η ημερήσια διάταξη τώρα προβλέπει τι δηλώσει του Συμβουλίου και τη Επιτροπή για την ανθρωπιστική κατάσταση των προσφύγων στα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να θυμίσω ότι μπορείτε να ζητήσετε να παρέμβετε βάσει τη διαδικασία ΚΑΤΣΤΙΑΗ και να χρησιμοποιήσετε την καλά σα κάρτα είτε με την κλασική μέθοδο εγγραφή είτε ηλεκτρονικώ. Να δοκιμάσετε και τα ηλεκτρονικά μέσα. Οι οδηγίε βρίσκονται στην, αίθουσα, στην είσοδο τη αίθουσα τη Ολομέλεια. Να δώσω τώρα το λόγο εκ μέρου του Συμβουλίου στην ε, Υπουργό Μπρνγκεκ. Και με συγχωρείτε αν προηγουμένω σα κατακρόκησα το επώνυμο. Αξιότιμοι βουλευτέ, για δεύτερη φορά επί της Προεδρίας μα είμαστε σε θέση να συζητήσουμε στην Ολομέλεια την ε, ανθρωπιστική κατάσταση σε σχέση με του πρόσφυγε στα σύνορα ε, αυτό σας ε, αποδεικνύει πόσο σημασία αποδίδεται και εμείς παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε όλους τους διαδρόμους ε, μετανάστευσης. Το 19 το σύνολο των παρανόμων διελεύσεων στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης υπολογίζεται στα 139.000 πρόσωπα ε, που ήταν 16% αύξηση σε σχέση με πέρσι και ε, όμως είμαστε στο κατώτερο ε, της εξαιτία όμως είχαμε 40% αύξηση των ανθρωπιστικών αναγκών και 60% σε σχέση με το 18% όσον αφορά τον διάδρομο Ανατολικής Μεσογείου όπου είχαμε διαλύσει πάνω 50% στα ελληνικά νησιά η κατάσταση προβληματίζει πάρα πολύ όπως όλοι είδαμε στην τελευταία συζήτηση που κάναμε εδώ στις 29 Ιανουαρίου. Ο αριθμός των προσώπων στα νησιά του Αιγείου έφτασε στο ρεκόρ ε, του να ξεπεράσει τα 40.000 πρόσωπα. Για πρώτη φορά έχουμε ε, το τόσο πολλά πρόσωπα κατά την εφαρμογή της συμφωνίας με την Τουρκία. Η Ελλάδα έχει λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να βελτιώσει τα πράγματα, ε, ανακοίνωσε νέα στρατηγική για προστασία των ανηλίκων που νομίμως διαμένουν στην Ελλάδα και ο στόχος είναι να ε, αυξηθεί η μεταφορά προσώπων στην κυρίω Ελλάδα. Ε, είχαμε πάνω από 35.000 που μεταφέρθηκαν στο παρελθόν. Συνεχίζεται αυτή η μεταφορά με αυξανόμενους ρυθμούς από την αρχή του 2020. Οι αφήξεις στην Ανατολική Μεσόγειο ε, έχουν επιπτώσεις άμεσες όσον αφορά τους μετανάστες και σε σχέση με την Ανατολική Ευρώπη. Είχαμε 14.000 παράνομες διελεύσεις ε, το 19 στα Δυτικά Βαλκάνια. Αυτό σημαίνει αύξηση 140% αύξηση σε σχέση με το 18. Από την αρχή του 20 η πίεση σε αυτό το διάβολο ε, αυξήθηκε, μειώθηκε λόγω του καιρού. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε μεγαλύτερη πίεση σε φετινό χειμώνα σχέση με τον προηγούμενο χειμώνα. Η Προεδρία θα συνεχίσει να προσέχει ιδιαίτερως το μεταναστευτικό, και θα αυξάνουμε τις δυνατότητες διαχείρισης στα Δυτικά Βαλκάνια. Θα προσέχουμε ιδίως το τι γίνεται σε Βοσνία Ζήγοβίνη για έχουμε προστασία των μεταναστών ε, και σύμφωνα με τον ΟΗΕ πάνω από 8.000 ε, μετανάστες πρόσφυγες υπάρχουν ε, κυρίως στα βορειοδυτικά σύνορα της χώρας. Η κατάσταση παραμένει προβληματική, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες είχαμε θετικές εξελίξεις, γιατί είχαμε ε, ε, βελτίωση στην υποδοχή. Ε, ο κύριος Μποζίνοβιτς, ο Υπουργός Ιστορικών, μίλησε με τον κύριο Ράντοσετς που είναι ο Υπουργός Ασφαλείας της Βοσνίας και συμφώνησαν να αναβαθμίσουν τη συνεργασία τους σε διάφορους σημαντικούς τομείς στην εφαρμογή μιας διαδικασίας επανεισδοχής για υποδοχής, να έχουμε μικτές περιπόλους στα σύνορα και βοήθεια προς την Κροατία όσον αφορά την ασφάλεια στα σημεία ελέγχου των συνόρων. Συμφώνησαν ναι, επίση να έχουμε καλύτερη συνεργασία όσον αφορά του, τα δίκτυα των λαδρεμπόρων και αυτό συζητήσει σε επίπεδο υπουργών σε μια άτυπη σύνοδο στο Ζάγκρεμπ στις 24 Ιανουαρίου του 20 από τους Υπουργούς Συνδικών της Ένωση. Ο Υπουργός ε, είπε ότι έχουμε τώρα ε, αύξηση των συνοριοφυλών κατά χίλιους στα σύνορα με τη Βοσνία και 93% αυξήθηκαν τα όσα δίνονται στην Βοσνία πέρσι για την ανθρωπιστική μεταχείριση των μεταναστών και 7% αφορούσε μόνο τη ε, τις δυνάμεις ασφαλείας. Θα συνεχίσει η Ένωση να βοηθά την Βοσνία, ούτως ώστε να υπάρχει εξοπλιστής μεταχείριση όλων των μεταναστών και κυρίως των πιο ευαλώτων ταυτόχρονα. Θέλουμε να υπάρχει μια λύση πιο διαρκής, πιο μόνιμη, πιο σφαιρική και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με όλους τους εμπλοκομένους στα Δυτικά Βαλκάνια και ο σκοπός ο απότερος είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι ροές αυτές στα σύνορά μας ε, έχουν σωστή διαχείριση, και πάντοτε γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα. Επίσης έχουμε αυτά τα πρόσφατα ελληνικά μέτρα που, ε, ότι θα βοηθήσουν. Η καινούργια νομοθεσία που τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα θα πρέπει να επιταχύνει τις εξελίξεις για επαναπατρισμούς και χορήγηση ασύλου. Είναι πολύ μικρές οι ροές επιστροφής για πολύ καιρό. Ε, θα πρέπει να γίνει διαχείριση των ροών και το σχέδιο της κυβέρνησης της Ελλάδος είναι η επιστροφή 10.000 μέχρι τέλος του 20. Ε, αυτό είναι φιλόδοξος στόχος, αλλά μπορεί να ε, γίνει εφικτός με βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πραγματικές αποτελεσματικές επιστροφές χρειάζονται όμως και συνεργασία της Τουρκίας. Για να εξασφαλίσουμε την χρηστή διαχείριση είναι σημαντικό οι εταίροι των Δυστικών Βαλκανίων να βελτιώσουν τις δυνατότητες διαχείρισης και στον τομέα των επαναπατρισμών αλλά και των εθελούσιων επαναπατρισμών να υπάρχουν ε, ε, επανεισδοχείς συμφωνίες με τις τρίτες χώρες ε, σύντονες με την πολιτική μας. Εμείς θα βοηθήσουμε προς όλες αυτές τις κατευθύνσεις όσο μπορούμε. Τώρα όσον αφορά το, το, τον διάδρομο της Κεντρικής Μεσογείου, τα πράγματα είναι χειρότερα στην Λιβύη γιατί υπάρχει ο εμφυλίος στη χώρα και για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ε, θυγέντες ε, μετανάστες και πρόσφυγες ε, τα κράτη-μέλη και η είπα αρμοστία του ΟΗΕ έχουν κάποια προγράμματα και κάποιο καταπίστευμα. Οπότε να γίνει διαχείριση των εθελουσίων επιστροφών και έτσι να υπάρχει ανθρωπιστική βοήθεια. Έγινε αυτό και οι επιδόσεις είναι σημαντικές. Ε, επίσης, ε, κάποιοι μεταφέρθηκαν σε Ρουάντα και από Ρουάντα Νίγηρα και πήγαν σε χώρες υποδοχής και στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την υποτερμοστία. Αυτό είναι σημαντικό γιατί ο φίλος του Λιβύης συνεχίζεται